αποτελεσματική στη δράση της, πάντως, έστω και την τελευταία στιγμή, εγκαίρως τουλάχιστον, ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Περατώθηκε αυτή η συζήτηση και τώρα στην εμμυρίσια διάταξη έχουμε την δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την κατάσταση στην Ιαπωνία, όπως επίσης και τον συναγερμό στους πυρηνικούς σταθμούς. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον, στην Υπουργό Γιώρη να μας μιλήσει εκ μέρους του Συμβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Ότεγκερ, οι βουλευτέ. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας ε, τα συλληπιτήριά μας προς τον λαό της Ιαπωνίας ε, για αυτούς που έχασαν τους αγαπημένους τους, τους και πολλούς άλλους που ε, επλήχθησαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από τα τραγικά περιστατικά πριν από δέκα ημέρες. Επίσης, να αποτίσω φόρο τιμή ε, στο κουράγιο και την αποφασιστικότητα αυτών που τώρα αγωνίζονται για να ανταπεξέλθουν με τις συνέπειες του φρικτού σεισμού και του τσινάμι, καθώς και όσους ε, ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τι συνέπειε των πυρηνικών περιστατικών η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι στο πλευρό των Ιαπώνων σε αυτή την εξαιρετική δύσκολη στιγμή. Έχουμε ήδη δώσει συγκεκριμένη βοήθεια στην Ιαπωνία. Την ίδια ημέρα που χτύπησε ο Αγγέλαδος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την υπάτη, από τον εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιήσει όλες όλα τα μέσα βοήθειας και κινητοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Πολιτικής Προστασίας για να δοθεί βοήθεια από τα κράτη-μέλη και εντός σύντομου χρονικού διάστηματος η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια της Ιαπωνικής κυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι, εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη για ανθρωπιστική βοήθεια, τεχνική αρρωγή ή οποιαδήποτε είδους ε, ειδικής βοήθειας που μπορεί να ζητήσουν οι Ιαπωνικές αρχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εξ ονόματος του Συμβουλίου την Επίτροπο Γεωργίευ και την ύπατη εκπρόσωπο που αντέδρασαν γρήγορα και συντονισμένα. Ε, η ομάδα πολιτικής προστασίας που έχει ε, δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία έχει την πλήρη υποστήριξή μας και τα μεμονωμένα κρατημέλη επίσης προετοιμάστηκαν να δώσουν βοήθεια. Είναι επίσης σημαντικό να κοιτάξουμε και το μακροοικονομικό αντίκτυπο της ιαπωνικής κρίσης. Οι υπουργοί είχαν μια προκαταρτική συζήτηση στο πλαίσιο του ΕΚΟΦΗΝ στις 15 Μαρτίου. Προφανώς, ένα από τα βασικά στοιχεία που μας ανησυχούν είναι η κατάσταση στο πρινικό σταθμό Φουκουσίμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ουγγρική Προεδρία έδρασε χωρίς καμία καθυστέρηση, λαμβάνοντα υπόψη τη σοβαρότητα τη κατάστασης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τον πυρηνικό κίνδυνο. Και ε, συγκλήθηκε κατευθείαν ε, η ομάδα εργασίας ατομικών ζητημάτων και ένα έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας για να αξιολογηθεί η κατάσταση στην Ιαπωνία και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το πρώτο μήνυμα του Συμβουλίου ήταν αλληλεγγύης ε, ε, και δημότητας για την παροχή ανθρωπιστικής και τεχνικής βοήθειας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα επίσης ε, σεβασμού για την ανθεκτικότητα και την επιμονή των Ιαπώνων, ιδιαίτερα όσων ε, αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν με την κατάσταση στην Φουκουσίμα. Χάρη σε αυτή την επιμονή βλέπουμε κάποια ελπίδα σε ό,τι αφορά την κατάσταση στις, ε, στα πυρηνικά εργοστάσια, στο εργοστάσιο, παρά το γεγονό ότι η κατάσταση παραμένει σοβαρή. Το βασικό πρόβλημα είναι τα υψηλά επίπεδα μόλυνση που έχουν μετρηθεί ε, κοντά στο σταθμό και πρέπει να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας προς την Ιαπωνία. Διάφορα κράτη-μέλη, είτε διμερός, είτε, μέρο, είτε μέσω διαφόρων μηχανισμών ε, συντονισμού, ε, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση ως ε, Επί του παρόντο, όπως είπε και ο Ούγκρο Υπουργό ε, Αγροτική ανάπτυξη δεν υπάρχουν επιπτώσει για τον ε, λαό τη Ευρώπη, για του λάου της Ευρώπης. Τα <clears throat> επίπεδα ε, ραδιενέργεια σε όλα τα κράτη-μέλη είναι κανονικά και συνεχίζονται οι έλεγχοι για τρόφιμα που εισάγονται από την Ιαπωνία. Ωστόσο, θα πρέπει να μάθουμε κάποια μαθήματα από το ατύχημα αυτό. Η συνεχιζόμενη εφαρμογή των υψηλών προτύπων ε, πυρηνική ασφάλεια αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φυσικά πρώτα θα πρέπει να εξαγάγουμε τα συμπεράσματα από το ατύχημα αυτό, παρά το γεγονό ότι δεν, ε, δεν προκλήθηκε από κάποια δυσλειτουργία στο εργοστάσιο, αλλά από εξωτερικού παράγοντε. Διάφορα κράτη-μέλη αποφάσισαν να αναθεωρήσουν την ασφάλεια των ε, πυρηνικών σταθμών τους, το οποίο και καλωσορίζουμε μετά το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στις 21 Μαρτίου. Ε, ο Υπουργό Φελέγγι ε, απέστειλε μια επιστολή προς τον Πρόεδρο Φαν για να προτείνει την διεξαγωγή stress test δοκιμών αντοχής και το εύρος εφαρμογής των δοκιμών αυτών θα πρέπει να αναπτυχθεί δεδομένων των πρόσφατων γεγονότων και της διαθέσιμης τεχνογνωσίας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το γεγονός επίσης ότι κάθε πυρηνικό εργοστάσιο έχει δικές του, δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κίνδυνο πλημμυρών, σεισμών ε, και σε ό,τι αφορά φυσικά και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η ομάδα, η ομάδα, Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Ομάδα Πυρηνικής Ασφάλειας με πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών θα ορίσει αυτούς τους παραμέτρους ε, για το, τη δοκιμασία, τις δοκιμές αυτές. Και θα πρέπει φυσικά να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν το θέμα της ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων. Ασφαλώς δεν ε, σταματάει στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συμμετάσχουν και οι γειτονικέ τρίτες χώρες. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών ε, εργοστασίων με την ε, πλήρη χρήση των διεθνών οργανώσεων και σωμάτων όπως ε, η Διεθνή Οργάνωση Πυρηνικής Ασφάλειας ή το G20. Είναι σημαντικό το ε, μήνυμά μας προς τον κόσμο δεδομένη της κατάστασης στην Ιαπωνία να είναι σαφές. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Καταρχάς, η αξιοπιστία του όλου εγχειρήματο στηρίζεται στην διαφάνεια του αποτελέσματος. Κατά δεύτερον, όσο και αν είναι σοβαρό το περιστατικό στην Ιαπωνία, δεν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας είναι κάτι που το εξετάζουμε για πρώτη φορά τώρα. Είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι υπάρχει δεσμευτικό νομικό πλαίσιο στην Ευρώπη εδώ και 25 χρόνια σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα πυρηνικά ζητήματα. Το Συμβούλιο ασφαλώς θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις και ε, εν πάση περιπτώσει θα εξετάσει το θέμα σε κάθε περίπτωση ότι και θα συμβεί τον Ιούνιο. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, στα τέλη τη εβδομάδα θα καταγράψει την κατάσταση στην Ιαπωνία μετά από την τραγωδία αυτή. Δεν αμφιβάλλω για το ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα εκφράσουν τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη του με τον λαό της Ιαπωνίας, όπως και κάνω και εγώ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι διαθέσιμη για να παράσχει οτιδήποτε βοήθεια χρειαστεί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και για μια φορά ακόμα θα ήθελα να χαιρετήσω το κουράγιο και την αποφασιστικότητά του. Σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο Επιτρόπος Ρετινιέρ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει τη σημασία της αλληλεγγύης με τον Ιαπωνικό λαό και την Ιαπωνική κυβέρνηση. Και έχουμε τονίσει τη συμπαράστασή μας με κάθε τρόπο. Έχουμε τονίσει και τη σημασία του θάρρους και της αυτοσυγκράτησης του Ιαπωνικού λαού. Έχουμε ξεκινήσει την συμβολή των κέντρων παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε δώσει αρρωγή με σκηνές, με στρώματα, με δοχεία για είδωρ, για υγειονομικό εξοπλισμό κτλ. Ήδη αυτές τις μέρες, την Πέμπτη το πρωί και την Παρασκευή, θα φτάσουν όλα αυτά τα αγαθά στην ε, Ιαπωνία και θα διανεμηθούν και η κυρία Επίτροπος Γεώργιεβα από την Κομισιόν θα είναι και υπεύθυνη για τα θέματα αυτά. Κάναμε επίσης προτάσεις προς την Ιαπωνία για βοήθεια στα πυρηνικά κέντρο και ε, αναμένουμε ακόμα την απάντηση της Ιαπωνικής πλευράς. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και παρακολουθούμε, αναλύουμε και αξιολογούμε την κατάσταση ασφαλείας στην Ιαπωνία. Για να μπορέσουμε να περατώσουμε την κατάσταση ανάγκης στους πυρηνικούς σταθμούς, αναμένουμε ότι οι Ιάπωνες τεχνικοί και μηχανικοί θα μπορέσουν να φέρουν σε πλήρη έλεγχο το πυρηνικό αυτό κέντρο και να αποφύγουν περαιτέρω ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να προξενηθούν στους αντιδραστήρες. Η Ευρώπη βέβαια πρέπει να αντλήσει κάποια συμπεράσματα από όλα αυτά τα στοιχεία. Έγινε ήδη μια συζήτηση με, τις, ε, με τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες που έχουν ρόλο στην παραγωγή ή στη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών και με τις υπηρεσίες εποπτείας για τους ατομικούς σταθμούς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κατών μελών. Και επίσης υπήρξε και μια έκτατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα θέματα τα, της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστό ότι είναι πολύ διαφορετικές οι θέσεις της, ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 17 χώρες έχουν πυρηνικούς σταθμούς και 13 από αυτά θέλουν να τα διατηρήσουν ως μόνιμο στοιχείο της ε, ενεργειακής τους πολιτικής. Η Γερμανία ίσως είναι μια εξαίρεση σε αυτά. <clears throat> Υπάρχουν δύο κράτη επίσης τα οποία έχουν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον την πυρηνική ενέργεια. <clears throat> Εκτός από τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες, τα θέματα επιλογής ενεργειακής ε, ε, ενεργειακού κράματος, ενεργειακής ε, επιλογής και ενεργειακού μείγματος είναι στην ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε, σε ορισμένες περιπτώσεις το μέσο όρος πυρηνικής ενέργειας είναι 30% στην Ευρώπη, αλλά είναι 8% μόνο στην Αυστρία και 80% στην Γαλλία. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη πολυπικιλία σε σχέση με τα θέματα αυτά και ανεξάρτητα από την τροπή που θα πάρει η κατεύθυνση της ποινική ενέργειας είναι σαφές ότι οι υποδομές για τη διανομή και την αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει να ενταθεί και να ενισχυθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Και έρχομαι επίσης και στο θέμα της ασφάλειας των σταθμών ενέργειας. Η ασφάλεια των σταθμών ενέργειας είναι πολύ σημαντική αλλά είναι ιδιαίτερο πρόβλημα και ιδιαίτερη μέρη να μα η ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, ώστε να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι σε αυτά και οι, Ευρωπαϊ... οι Ευρωπαίοι πολίτες και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η πρότασή μας λοιπόν βρίσκεται τώρα υπό επεξεργασία για το κατά πόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από τα γεγονότα της Ιαπωνίας, τα φαινόμενα τα οποία αναγνωρίσαμε επομένως στην πυρηνική αυτή καταστροφή και να δούμε κατά πόσον θα πρέπει στην Ευρώπη να εφαρμόσουμε κοινά πρότυπα με στόχο μια μείωση των κινδύνων ώστε τα 130 περίπου ποινικά εργοστάσια τα οποία βρίσκονται στην Ευρώπη να εξασφαλιστεί η ασφαλειά τους και ώστε να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα για τα νέα πυρηνικά εργοστάσια τα οποία δύναται να δημιουργηθούν στην Ευρώπη ανεξάρτητα λοιπόν για το αν ένα κράτο μέλο θέλει να διατηρήσει την πυρηνική ενέργεια, να χρησιμοποιήσει το μέλλον που δεν τη χρησιμοποιεί τώρα ή να φύγει από την πυρηνική ενέργεια, θα πρέπει να έχουμε κοινά κριτήρια για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε θέματα όπω πλημμύρε, όπω ε, σεισμοί, τα προβλήματα τα οποία μπορούν, όπω είδαμε στην Ιαπωνία, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα των ε, συστημάτων ψήξεως τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε ε, ηλεκτρικό ρεύμα με πρόσθετους εξοπλισμούς στους πυρηνικούς σταθμούς ώστε να αντιμετωπίσουν τα επακόλουθα πλημμυρών ή σεισμών. Ο στόχος μας είναι να έχουμε και συγκεκριμένες προδιαγραφές για τους ποινικούς σταθμούς ανάλογα με την ηλικία τους, με την τεχνολογία τους, με το σημείο στο οποίο έχουν κατασκευαστεί, τη σεισμικότητα κτλ. Επίσης, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πτώσεις αεροσκάφου σε ποινικούς σταθμούς, κυβερνοεπιθέσεις, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κοινή αυτή εξέταση των ποινικών σταθμών. Θέλουμε να έχουμε μια επιτροπή η οποία θα προετοιμάσει τα θέματα αυτά μαζί με τις υπηρεσίες ατομικής ενέργειας τα κράτη-μέλη φυσικά έχουν την ευθύνη για τα θέματα αυτά, αλλά μπορούν εθελοντικά να δεχτούν να υποβληθούν σε ένα κοινό stress test για τους πυρηνικούς σταθμούς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Πρόεδρος Συμβουλίου μίλησε και για γειτονικέ χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικούς σταθμούς και μπορεί αυτό να έχει επίπτωση στην ασφαλεία μας. Ουκρανία, Αρμενία, Τουρκία, Ρωσική Ομοσπονδία είχα μια μακρά τηλεφωνική επαφή με τον Υπουργό Ενέργειας της ε, Ουκρανίας τόνισα ότι μπορεί να συμμετάσχει στο κοινό στρες τεστ των πυρηνικών σταθμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, εμείς είμαστε αρμόδιοι για τα τεστ αυτά έναντι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την ενότητα αυτών των στρες τεστ. Εάν δεν θέλει ένα κράτος μέλος να συμμετάσχει σε αυτά, τότε φυσικά μειώνεται και το κύρος που έχει η πρότασή μας έναντι γειτονικών χωρών όπως είναι η Τουρκία, η Ουκρανία, η Ελβετία κτλ. Στις επόμενες λοιπόν εβδομάδες θα πρέπει να προετοιμαστούν τα κριτήρια ασφαλείας και είμαι απόλυτα διαθέσιμος να συζητήσω αυτά τα κριτήρια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με όλους τους εμπλεκομένους, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, επιχειρήσεις ενέργειας, ενώσεις επιστημόνων και τεχνικών. Να συνεργαστούμε λοιπόν με όλους αυτούς με το στόχο να έχουμε ένα όσο το δυνατότερο πληρέστερο πλαίσιο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα ασφαλείας και να αυξήσουμε το επίπεδο ασφάλειας και πρόβληψης για τα θέματα αυτά. Ο στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε μια γενικότερη απόφαση σε επίπεδο των G20, όχι μόνο για τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχατε, είδατε ήδη ότι εγώ ήμουν παρόν και στην Επιτροπή Ενέργειας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά, ζητώντας την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι θα έχω αύριο και αντίστοιχη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπη. Τώρα ε, θα μιλήσουν οι πρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Αρχίζουμε με την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο κύριος Μπροκ, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επιτροπή, συνάδελφοι. Νομίζω ότι η ισχύ της φύσεως ε, ε μας έγινε και πάλι σαφής και βλέπουμε τα όρια της ανθρώπινης ε, ικανότητης και το πόσο παραδομένοι είμαστε ε, έναντι της βίας της ε, φύσης. Σε τέτοιες στιγμές δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη μας με την Ιαπωνία. Αλληλεγγύη η οποία εκφράζεται και με σκέψη και με προσευχή αλλά και με πρακτική βοήθεια και όπως είπε ο Επίτροπος η παροχή βοήθειας ε, έχει ως σκοπό να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε, να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε και ξέρω ότι δεν είναι μόνο οι κρατικές δομές αλλά και πολλοί πολίτες που στην Ευρώπη είναι δεθυμένοι να δώσουν χρήματα. Στην ε, Γερμανία μας συλλέχθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες 50.000 ε, ευρώ και συνεχίζονται οι ενέργειες αυτές. Παράλληλα θα πρέπει να προσέξουμε να μην χρησιμοποιηθεί αυτό για εσωπολιτικά ζητήματα. Θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από το πυρηνικό ατύχημα να διεξάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα stress test γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν σύνορα σε περιπτώσεις τέτοιων ατυχημάτων και να κοιτάξουμε να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τα υφιστάμενα εργοστάσια, για την υφιστάμενη τεχνολογία. Μιλήσαμε και για αλλαγή κλίματος, για απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Αλλά κυρίες και κύριοι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και ο όρος υπόλοιπη κίνδυνη θα οριστεί καλύτερα. Η Ιαπωνία θα αλλάξει τον τρόπο, μας, τον τρόπο σκέψης μας, την οτροπία μας ε, σε αυτή την άποψη. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο, ο εναπομείνοντας κίνδυνος θα πρέπει να συνεπάγεται μια αλλαγή σκέψης και μια αλλαγή πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θεωρώ αυτό αναγκαίο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. η κυρία Ουλσκοβ, δύο λεπτά. Πρόεδρε. Μία από τις πιο αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την τεχνολογική και την οικονομική ε, ζωή έχει καταρακωθεί από την καταστροφή αυτή. Φυσικά οι πρώτες σκέψεις μας ε, πάνε στους ανθρώπους και οι εικόνες που βλέπουμε καταδεικνύουν την κατάσταση και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, αλλά βλέπουμε πόσο ευάλωτη είναι όλη η κοινωνία. Αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία θα μπορούσε να συμβεί σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και εδώ, ακόμα και σε χώρες που έχουν υψηλά πρότυπα ασφάλεια. Φυσικά, αναγνωρίσουμε τα θέματα πρινικής ενέργειας. Κοιτάξτε, κάποιες χώρες δεν έχουν πρινική ενέργεια, αλλά κάποιες άλλες εξαρτώνται πολύ από τα πρινικά εργοστάσια. Κάποιες χώρες φτιάχνουν καινούργια εργοστάσια, αλλά σκοπεύουν να τα καταργήσουν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά και διαφορετικά επίπεδα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που παράγουμε ενέργεια για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τους κινδύνους. Για να αυξήσουμε την άμυνά μας θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη προκειμένου μακροπρόθεσμα να χρησιμοποιηθούν πηγές ε, ανανεώσιμης ενέργειας. Είναι τεράστιο το δυναμικό που μας ε, παρέχουν αυτές οι μορφές ενέργειας. Σε αντίθεση με την οικοδόμηση νέων εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας, οι οποίες απλά θα συνεχίσουν, να μας, ε, θα συνεχίσουν την εξάρτηση από αυτή την ε, πηγή ενέργειας. Γιατί να μην ξεκινήσουμε λοιπόν από σήμερα. Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς μπορούν να θεθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο υψηλή στόχοι σε ό,τι αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και για το πώς μπορεί να καταστεί η ανανεώσιμη ενέργεια τμήμα του ενεργειακού μείγματος και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν έτσι, δοκιμές αντοχής σε όλα τα πρινικά εργοστάσια στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε για το μάτι των ελευθερών, η κυρία Εκ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η εικόνα του μεγάλου σεισμού και του τσουνάμι στην βορειοανατολική Ιαπωνία δημιουργούν φρίκε και η σκέψη μας πάνω σε αυτούς που χάσανε τους δικούς τους, τα σπίτια τους, και να επικροτούμε το πακέτο της Ένωσης. Στη Φουκουσίμα ακόμα το προσωπικό δουλεύει στους πυρηνικούς σταθμούς προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω ρήπανση λόγω ακτινοβολίας. Και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί με πάρα πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο από όλη την Ένωση και στις Βρυξέλλες. Επικροτώ τα, τα τεστ που πρότεινε η Κομισιόν. Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σε τεστ όπως της ε, γεωγραφίας και τεχνολογίας. Χρησιμοποιούμε σε άλλα δύο τεινά. Το ένα είναι μια κουλτούρα ασφάλειας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε βέβαια τους πολλαπλούς κινδύνους, ενώ το κάνουμε αυτό. Και το άλλο είναι το θεσμικό πλαίσιο. Μια εποπτεία και των σχέσεων μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών οργάνων και των εταιριών που ασχολούνται με τα πυρηνικά οι αρχές δεν θα πρέπει να τους επιτρέπουν να αυτοελέγχονται. Τέλος, να αξιολογήσουμε τις συνέπειες της καταστροφής με συζήτηση με βάση πληροφορίες και γνώση. Ίσως χρειαστούν ριζοσπαστικά μέτρα. Απαιτούνται μάλλον μέτρα, αλλά ένα είναι δεδομένο. Ότι πρέπει να μετερρυθμίσουμε την παραγωγή ενέργειά μας για να στηριζόμαστε περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Για την ομάδα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, ο κύριος Τσίτσεστερ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω το θαυμασμό μου για την στοική ανθεκτικότητα που έδειξε ο Ιαπωνικός λαός εν ώψη της βίαιης καταστροφής που υπέστη από τις δάμεις της φύσης. Πρέπει να θυμόμαστε πόσο έντονος ήταν ο σεισμός και το τσουνάμι. Εγώ χαιρετίζω τα προληπτικά stress για τους ε, ευρωπαϊκούς πυρηνικούς σταθμούς. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η πυρηνική βιομηχανία είναι ήδη η πιο υποκείμενη σε ρύθμιση και η πιο ενεπιγνώση των κινδύνων σε όλο τον κόσμο. Και φέτος η Μπένρο, η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών Πυρηνικών Σταθμών, έκανε προτάσεις για να γίνουν οι νέοι πυρηνικοί σταθμοί ακόμα και πιο ασφαλείς από τους τωρινούς. Πρέπει να συγκρίνει κανείς την ε, ασφάλεια, το ιστορικό ασφάλεια των υδροηλεκτρικών, θερμικών και άλλων σταθμών με την πυρηνική βιομηχανία σε σχέση με απώλεια ζωής. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να έχουν και μια θετική πτυχή η καταστροφή της Ιαπωνίας. Ότι η ανοικοδόμηση της χώρας αυτής με την υποστήριξη των ασφαλιστικών εταιριών θα πρέπει να δώσει μια ισχυρή όθηση στην οικονομία της Ιαπωνίας και αυτό θα είναι θετικό για όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο, την κυρία Υπουργό και τον κύριο Επίτροπο για αυτά τα οποία είπαν και θέλω να πω στα κράτη-μέλη να μην χάσετε το θάρρος σας για την πυρηνική ενέργεια. Τώρα εξακολουθούμε να τη χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πράσινους η κυρία Χάρμς για τρία λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εννοείται ότι σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Ιαπωνία όσο καλύτερα μπορούμε και με οποιαδήποτε μέσο έχουμε στη διάθεσή μας ε, σε μια χώρα η οποία έχει πληχθεί από μια τέτοια καταστροφή χρειάζεται κάθε βοήθεια αλλά θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτο το πόσο εύκολα ε, μιλάμε και επενούμε τους ήρωες στην Ιαπωνία. Δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτοί που αποκαλούμε ήρωες, αυτοί ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον ότι παίζουν τη ζωή τους ε, και αυτοί που καταπολεμούν την πυρηνική καταστροφή στην Φουκουσίμα απειλούνται από θάνατο. Κανένας λαός δεν ξέρει σε όλο τον κόσμο τόσο καλά τι σημαίνει και τι μπορεί να κάνει μια πρινική καταστροφή από την Ιαπωνία. Έχει σημαντευτεί η ιστορία τους από τη Χρυσή Αγκασάκη. Κάθε παιδί ξέρει ποιε είναι οι συνέπειες μιας πρινικής σύνθηξης. Αυτό να το αντιληφθούμε, να το συμμετοποιήσουμε όταν μιλάμε για την Ιαπωνία. Ο τρόμος, ο οποίος δεν έγινε μόνο στη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά και θα ακολουθήσει στο μέλλον, στο μέλλον είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν οι Ιάπωνες καλύτερα από κάθε άλλον. Ίσως και οι Ουκρανοί να μπορούν που γνωρίζουν ένα τμήμα της κόρης τους ως απεριμωμένο τμήμα. Ίσως αυτοί μπορούν να μιλήσουν επίσης. Ε, στην ευρωπαϊκή συζήτηση το θέμα θεωρώ είναι το εξής. Δεν είναι το ίδιο όπως πριν από 25 χρόνια. Δεν είναι το θέμα να συζητήσουμε τις συνέπειες, τις πολιτικές συνέπειες όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια τεχνολογία στις χώρες μας η οποία σε περίπτωση αμφιβολίας μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και όχι μόνο να καταστρέψει και το παρελθόν και το παρόν αλλά και το μέλλον μιας περιοχής, το μέλλον όλων που ζουν στην περιοχή αυτή αλλά και στην ευρύτερη, στο ευρύτερο κοντινό περιβάλλον. Δεν Νομίζω ότι έχει νόημα να μιλάμε για δοκιμέ ε, αντοχή κυρία Ότιγκερ, να είμαστε πιο ειλικρινεί. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά στα εργοστάσια μα, αντιμετωπίζουμε καταστάσει που είναι κοντά σε πυρηνική σύνταξη. Να σα πω ότι αν στο Βέλγιο, στη Βόρεια στην Γαλλία, Φίλιξμπουργκ στη Γερμανία, ή στη Βουλγαρία, Πάξ στην Ουγγαρία, Προυσπίτελ με έκρηξη υδρογόνου στην ε, Γερμανία. Μπάζοβικ στη Σουηδία, στη Γερμανία, στην Γαλλία. Μιλάμε για τα πιο εντυπωσιακά ε, παραδείγματα, τα οποία ε, έχουμε πλησιάσει μάλλον πιο πολύ από κάθε άλλη φορά μετά το Τσέρνομπιλ σε πυρηνική σύνδεξη. Πώς ε, θα καταφέρουμε σε κάθε, πυρηνική, σε κάθε πυρηνικό εργοστάσιο Μάλλον πώς ε, συμβαίνει αυτό, να έχουμε πλησιάσει τέτοια περιστατικά σε όλα τα πυρηνικά εργοστάσια. Τα stress έχουν ε, κάποιο νόημα αν οδηγήσουν σε κάποιο σχέδιο για το ποια εργοστάσια, ποια κέντρα θα πάψουν να λειτουργούν. Αν ε, τα τεστ αυτά τελικά ε, μας οδηγήσουν στην Ευρώπη στο να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Ιαπωνία. Και θα συζητήσουμε επίσης ποιος θα κάνει, ποιος θα ορίσει τα, τις δοκιμές αντοχής. Δεν μπορούν να είναι αυτοί οι διευθυντές, οι διαχειριστές, οι διοκτήτες των πυρηνικών εργοστασίων και ποιος θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα. Γιατί ως τώρα ε, κλείναμε τα μάτια της, ε, ενώπιον των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Και πολύ συχνά η Euratom, στην περίπτωση του Μόχοφτσα για παράδειγμα, ενέκριναν εργοστάσια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα, έπρεπε να έχουν λάβει έγκριση. Σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας για την ε, ομάδα της ε, Ενωμένης Αριστεράς, ε, κυρία Ντεμπρούν. Ένα λεπτό. Θα ήθελα να προσφέρω τα συλληπιτήριά μου προς αυτούς που επιλήγησαν από την τραγωδία στην Ιαπωνία, μια τραγωδία που συνεχίζεται. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε το λαό της Ιαπωνίας από τα μαθήματα που έχουμε να δεθούμε στην Ευρώπη το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας είναι στην ημερήσια διάταξη πια σταθερά ιδιαίτερα όσον αφορά τα τεστ κόπωσης που πρέπει να γίνουν στους πυρηνικούς σταθμούς της Ευρώπης. Δεδομένου αυτού που συνέβη στην Ιαπωνία υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Η ανθρώπινη τραγωδία δείχνει την ανάγκη να περάσουμε σε μια μη πυρηνική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα μορατόριο για την πυρηνική ενέργεια και χρειαζόμαστε και πολλές επενδύσεις σε ενέργεια που να είναι βιώσιμη και ανανεώσιμη πρέπει να γίνει αναθεώρηση του ρυθμιστικού επίσης συστήματος όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ για την ομάδα Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ο κύριος Προβέρα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια, το σθένος που επέδειξε ο Ιαπωνικός λαός μπροστά σε μια τραγωδία που σπάνια συμβαίνει στον κόσμο σε τέτοιες διαστάσεις. Η συμπεριφορά του Ιαπωνικού λαού πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους μας και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Το δίδαγμα που πρέπει να βγάλουμε από την εμπειρία αυτή είναι η ανάγκη να ενισχυθεί το σύστημα προστασίας του πληθυσμού στην Ευρώπη με πιο αυστηρό συντονισμό των παρεμβάσεων και να υπάρχει καλύτερη χρήση μέσων και ανθρώπων για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα σε περίπτωση καταστροφής. Όσον αφορά την επιλογή της πυρηνικής ενέργειας, το να συζητάμε σήμερα με βάση το, το τι συμβαίνει σήμερα θα ήταν λάθος, γιατί το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιστημονικά. Είναι πολύ σωστό ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα ασφάλειας για τους πυρηνικούς σταθμούς σήμερα και τη νέα γενιά, και να αποδομήσουμε του πιο παλιούς που είναι λιγότερο ασφαλεί. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε πολιτικές σκοπιμότητες, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και συνετοί όπω είπε ο συνάδελφο Μπροκ. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Φουκουσίμα, στο σεισμό, κατέβησε και ένα φράγμα με πάρα πολλά θύματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε όλα τα φράγματα ή δεν θα κάνουμε νέα φράγματα. Σύνεση λοιπόν, προσοχή και άνοιγμα όσον αφορά το μέλλον. Πρόεδρο, Ευχαριστούμε πολύ. Για τους μη ο κύριος Γκόλινης. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, η τρομερή καταστροφή που κτύπησε την Ιαπωνία, την βορειοανατολική Ιαπωνία, φυσικά προκαλεί την, ε, τη συμπαράσταση και τη συμπάθεια όλων των Ευρωπαίων που έχουν ε, κλονιστεί από αυτά τα γεγονότα. Πρέπει προφανώς να συμμετάσχουμε στις ενέργειες ανακουφιστικού Τη ενέργειας γιατί η κατάσταση δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί. Στην Ιαπωνία, κάθε άλλο, είναι μια χώρα η οποία έχει απόλυτη αίσθηση καθήκοντος αλλά όπου η γραφειοκρατία μπορεί να παραλύσει τις απαραίτητες ενέργειες. Έδειξε αυτή η κρίση ότι η βοήθεια που έρχεται από τη θάλασσα είναι πιο αποτελεσματική, αλλά φυσικά θα πρέπει να έχει κανείς και επαρκείς πλατφόρμες για την εκφόρτωση. Η κατάσταση δεν έχει βέβαια σταθεροποιηθεί ακόμα στην Ιαπωνία και είναι πολλοί οι οποίοι έχουν φύγει από τις αιστείες τους που έχουν πληγεί από την πείνα και από το ψύχος. Τα διδάγματα τώρα αυτής της τραγωδίας κατά την άποψή μου είναι τα εξή. Πρώτα απ' όλα ότι το χειρότερο πάντα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο Τιτανικός είχε κατασκευαστεί σαν ένα πλοίο το οποίο δεν μπορούσε να βουλιάξει. Ούτε ο Θεός δεν μπορούσε να το βουλιάξει, λέγανε. Αυτή ήταν η, η διαφήμιση αυτού του πλοίου. Και τελικά παρά τα στεγανά του διαμερίσματα, κατάφερε να βουλιάξει στο πρώτο του ταξίδι, γιατί δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι το χτύπημα του παγόβουνου μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη έκταση. Και το χειρότερο έγινε στην Ιαπωνία. Ο σεισμός μαζί με το τσουνάμι ήταν το χειρότερο δυνατό, ε, το χειρότερο σενάριο. Μπορεί να γίνει στην Καλιφόρνια, στην Κατώνα, στην Ιταλία, στην Καραϊβική ένας μεγάλος σεισμός αντίστοιχης έντασης Όλα αυτά πρέπει να τα προβλέψουμε λοιπόν με μια ενίσχυση τη πολιτική προστασία. Και το τελευταίο δίδαγμα είναι ότι παρόλα αυτά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Θα πρέπει, <clears throat> δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δεχόμαστε την πυρηνική ενέργεια ενώπιον του κινδύνου και συγχρόνως ότι δεν μπορούμε να έχουμε την ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα λόγω των αποβλήτων. Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι ομιλητέ, ξεκινώντα με την κυρία Καλνιέτε για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τραγωδία που έχει πλήξει την Ιαπωνία είναι πράγματι τρομερή. Εγώ θέλω να εκφράσω τα βαθιά συλληπιτήριά μου σε όλους αυτούς που επλήγησαν από την τραγωδία και στις οικογένειες των οικείων τους. Εγώ έχω θαυμάσει ιδιαίτερα την αυτοσυγκράτηση και το θάρρος που έδειξαν οι Ιάπωνες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και μπορούμε όλοι να πάρουμε διδάγματα από αυτούς. Η Ιαπωνία έχει τώρα να αντιμετωπίσει ένα έντονο έργο ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν. Αυτό θα χρειαστεί πολλά κονδύλια και μεταξύ αυτών και επενδύσεις από έξω από την Ιαπωνία. Στην συνάντηση κορυφή με την Ιαπωνία που θα γίνει στι 25 Μαου, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία. Αυτή η συμφωνία πρέπει να είναι ευνοϊκή και για τι δύο πλευρέ. Θα πρέπει να εξασφαλίσει μια ισοδίκαια πρόσβαση και στι δύο πλευρέ σε ό,τι αφορά τα βασικά προϊόντα, τι υπηρεσίε αλλά και τα αγροτικά προϊόντα. Μια τέτοια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσει το άνοιγμα των εμπορικών σχέσεων με την ε, Ιαπωνία. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα από το τσουνάμι είναι κάτι που έχει απασχολήσει <clears throat> και ανησυχήσει όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στους ηρωικούς ε, εργαζόμενους που ακόμα και τώρα διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στη Φουκουσίμα. Η εμπειρία όμως που έχουμε αποκομίσει από αυτήν την ε, καταστροφή, ιδίω από την πλευρά των Ιαπώνων τεχνικών και επιστημόνων, είναι μοναδική. Πρέπει να την χρησιμοποιήσει όλος ο κόσμος. Το γεγονός που έλαβε χώρα στη Φουκουσίμα θα πρέπει να οδηγήσει σε μία μίζωνα επιχείρηση δοκιμασίας των πυρηνικών σταθμών σε όλο τον κόσμο και για τη βελτίωση των πυρηνικών προτίμων. Και κλείνοντας θέλω να πω και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατό, ό,τι περνάει από το χέρι για να βοηθήσουμε την Ιαπωνία που είναι ένας από τους στενότερους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Childers, για ένα μισή λεπτό. Κυρία Childers. Κυρία Πρόεδρε, δύο πράγματα βγήκανε από το... τις μέρες αμέσως μετά τον τραγικό σεισμό στην Ιαπωνία. Πρώτον, η Ιαπωνέζικη αντίδραση γρήγορη η κινητοποίηση των μονάδων επίγουσα ανάγκη και το, η, ευελιξία που επέδειξε ο ιαπωνικό λαό. παραδειγματικά και θα πρέπει να είναι ε, παράδειγμα και για άλλε χώρε που γίνονται από σεισμού. Όμως η δεύτερη περίπτωση, το πυρηνικό ατύχημα στη είναι πιο δύσκολο. Η Ιαπωνία αναφεσβήτητα γρήγορα θα διδαχθεί από τα γεγονότα αυτά, αλλά και η Ευρώπη θα πρέπει να διδαχθεί. Και η αντίδρασή μα θα πρέπει να στραφεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών που λειτουργούν στην Ένωση. Τα τεστ ευπρόσδεκτα. Αλλά πρέπει να έχουμε κοινού κανόνε μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών και για την αποθήκευση υψηλά δραδιενεργού υλικού. Αυτό αφορά την Ιρλανδία, την εκλογική μου περιφέρεια, όπου υπάρχει πάρα πάρα πολύ υλικό που το κρατάνε στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Σέλαφιλ στην Αγγλία 280 χιλιόμετρα απόσταση από το κάντι ντάρον της περιοχής μου δηλαδή. Το δεύτερο είναι το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Χρειάζεται να σταματήσουν εντελώς η κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών. Για να συνεχιστεί να έχουμε επαρκή παροχή ενέργειας στην Ένωση χρειάζονται επενδύσεις σε ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και καλύτερη εξοικονόμηση της ενέργειας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Βαν Μπάλεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύμφωνα με τους συναδέλφους σε ό,τι αφορά τον σεβασμό προς τους ε, Ιάπωνες και το ότι συμπάσχουμε μαζί τους. Ωστόσο θα πρέπει να διδαχτούμε και αυτό τι σημαίνει ότι η καταστροφή αυτή η ενδυνάμει πυρηνική καταστροφή θα πρέπει να έχει και να λάβει μια διεθνή διάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Και για το ότι δεν δόθηκε συνέχεια στην ειδοποίηση, δεν συζητήθηκε η ειδοποίηση της Διεθνούς Οργάνωσης Πυρηνικής Ενέργειας. Θα πρέπει να μάθουμε τι συνέβη. Συμφωνώ με όλους όσοι είπαν ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουμε για την ανοικοδόμηση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική μια συμφωνία ε, ζώνης ελευθέρου εμπορίου και γι' αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριος Πιετρόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ως μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ω μέλο τη αντιπροσωπεία για τι σχέσει με την Ιαπωνία θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και να εκφράσω και την αλληλεγγύη μου προ το λαό τη Ιαπωνία ε, για την καταστροφή που κόστησε τη ζωή σε δεκάδε χιλιάδε ε, ανθρώπους, ενώ αγνοούμενοι εξακολουθούν να είναι 6.000 άτομα άνθρωποι. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία αλλάζουν ακόμα και είναι και τεράστιες και ηλικές ζημιές. 300 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι είναι οι ζημιές. Η, Ευρωπαϊκή, η, η Ιαπωνία δεν έχει στραφεί για βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραμείνουμε παθητικοί εν ώψη της τραγωδίας αυτής και κυρίως ανησυχούμε για την κατάσταση στο πυρηνικό σταθμό της Φοκουσίμα. Υπολογίζονται ότι θα είναι αντίστοιχο ο αντίκτυπο με αυτόν του Τσέρνομπιλ και θα πρέπει να μεταβούν εμπειρογνώμονε στην Ιαπωνία και να διαβουλευτούν με την κυβέρνηση της Ιαπωνίας προτού ξεκινήσουν οι... Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο ο κύριο Τούρμες. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι εταιρείες οι Ιαπωνέζικες οι οποίες δημιούργησαν τα πυρηνικά εργοστάσια στη Φουκουσίμα όπως είναι το ΣΥΜΠΑ είχαν πει πριν από στις μπροσούρες που δημοσιεύαν ότι είχαν τους πιο ασφαλείς ε, αντιδραστήρες στον κόσμο. Πιστεύω ότι η πάρα πολύ σοβαρή και θλιβερή καταστροφή που έλαβε χώρα θα πρέπει να δείξει και στην Ιαπωνία ότι δεν έχει κανένα νόημα, ότι είναι παράλογο να θέσουμε εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ένα πυρηνικό σταθμό έναντι ενός σταθμού ε, αιωλικής ή ηλιακής ενέργειας. Αυτή η ιδέα ότι είναι ανανεώσιμη η πυρηνική ενέργεια είναι λαθασμένη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει σε όλες τις μορφές ενέργειας. Και αυτό είναι το πρώτο δίδαγμα, κύριε Έτογκερ. Μήπως στον οδικό χάρτη για, μέχρι το 2050 να έχετε ένα σενάριο μέσα στο οποίο να προβλέπετε η χρησιμοποίηση το, από το 2050 και μετά 100% ανανεώσιμης ενέργειας. Για τα stress test εμείς τα υποστηρίζουμε. Αλλά θα πρέπει να έχουν ένα υποχρεωτικό χαρακτήρα και όχι μονάχα ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Τα stress test για τις τράπεζες ουσιαστικά είχαν χειραγώγησης από τις εθνικές αρχές και μόνο τη δεύτερη φορά άρχισαν να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα δεύτερο στοιχείο που απαιτείται είναι ανεξάρτητη ε, εμπειρογνωμοσύνη. Όταν έχουμε εταιρείε όπως η Aeon, Fantaisen λοιπά, οι οποίοι είναι οι εμπειρογνώμονες για τα θέματα πυρηνικής ενέργειας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, υπάρχουν πάντα εκπρόσωποι αυτών των εταιριών. Ακόμα και οι εθνικοί υπάλληλοι ξέρουν και μπορούν να το αποδεχτούν ότι οι έλεγχοι που έγιναν πριν από έξι μήνες δεν έχουν πια αγκυρότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν πραγματικά ανεξάρτητους εμπειρογνώμους για να κάνουν αυτές τις ε, αυτές, αυτούς τους ελέγχους. Και κύριε Εωτήγκερ ήμουν προσεκτικό δεν ανέφερα σε αυτά που είχε πει ο κύριος Σαρκοζή, ο οποίος είναι μεγάλος υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βίλς για ένα λεπτό έχει το λόγο. Στην Ιαπωνία εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος του μεγαλύτερου δυνατού πυρηνικού ατυχήματος. Ανεβαίνει ακόμα η ρεδιενέργεια στην ε, Φουκουσίμα και φάνηκε και πάλι με ένα τρομερό τρόπο ότι δεν μπορούν να είναι ελέγξιμοι οι πυρηνικοί σταθμοί. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε από την πυρηνική ενέργεια η οποία εξυπηρετεί μονάχα τα κέρδη των εταιριών ε, ενέργειας ενώ τον κίνδυνο ενό ατυχήματο θα πρέπει να τον επομιστούν οι πολίτες και οι καταναλωτές. Λοιπόν πρέπει να έχουμε επομένω μια σειρά προδιαγραφών η οποία να προβλέπει όλες τις καταστάσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν και να δημιουργήσουν ζημίες για τους πολίτες και το περιβάλλον. Θα πρέπει να φύγει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτά τα οποία διεκδικούν οι εταιρείε ποινική ενέργεια και να σταματήσει τη χρήση τη ποινική ενέργεια. Δεν μπορούμε να δίδουμε χρήματα των φορολογούμενων για μια τόσο επικίνδυνη μορφή ενέργεια όταν υποχρηματοδοτούνται όλε τι προσπάθειε για τι ανανεώσιμε ενέργειε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μάουρο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήταν σοβαρό λάθος νομίζω να μετατρέψουμε αυτή τη συζήτηση σε ένα είδος δίκη κατά των κινδύνων του εξυγχρονισμού. Η επιστήμη και η τεχνολογία μας επιτρέπουν να ζούμε περισσότερο, να ζούμε καλύτερα, να ζούμε με περισσότερο εμπιστοσύνη, διότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες της επιστημιστικής ασφάλειας, των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκε ενός κόσμου ο οποίος κοιτάει προς το μέλλον. Χωρίς τεχνολογία δεν θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Βέβαια, κίνδυνοι υπάρχουν. Και οι κίνδυνοι αυτοί είναι υπερβάσιμοι αν ξέρουμε να τους αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα που καθημερινά τίθενται στη διεθνή κοινότητα. Ιδιαίτερα σωστά είπε ο Έλμερ Μπρόκ. Υπάρχει ένα μυστήριο στη σχέση μας με τα πράγματα που μας κάνουν καταλάβουμε ότι δεν είμαστε κύριοι των πάντων. Έχουμε προχωρήσει αρκετά, αλλά δεν έχουμε απάντηση σε όλα τα προβλήματα που θέτει η φύση στον άνθρωπο. Και ο σεισμός αυτός ακριβώς μας θυμίζει ότι πιθανότατα συνθήκες κατώτερης τεχνολογίας πρόσφατα ή πριν από 100 χρόνια έδωσαν 100.000 νεκρούς στη Μεσίνα με πολύ λιγότερα ρίχτερ. Αυτά μας είναι χρήσιμα για το μέλλον. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι εργαλεία. Πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε μια σωστή πολιτική. Σωστή πολιτική αυτό είναι που θα κάνουμε από κοινού. Να βρούμε λύσεις για να ξεπεράσουμε την ατομική εποχή και να προβληθούμε στο μέλλον ή αν θα πρέπει για καιρό ακόμα να συζητάμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Σήμερα υπάρχει κάτι επομένο να κινητοποιηθούμε ειδικά για τον πόνο και τις ανάγκες ενός λαού. Δεν άκουσα πολλά λόγια γι' αυτό εδώ μέσα. Όλοι μας προβληματίζει και μας απασχολεί μια πολιτική συζήτηση που θα ξεκινήσει. Και ξεχνάμε πράγματα που έχουν άμεση σχέση με την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο, η κυρία Σάρμπου, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κρίση στην Ιαπωνία μας ανησυχεί όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών σε όλο τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι να μας θέσουμε το ερώτημα η πυρηνική μας σταθμή είναι ανθεκτική, είναι ασφαλής. Εγώ προέρχομαι από τη Ρουμανία και οι συμπολίτε μου ανησυχούν όσον αφορά το σταθμό της Τσερναβόντα κυρίως διότι στον τύπο υπάρχουν άρθρα που βάζουν και ερωτηματικά και θαυμαστικά. Και δεν είναι κατάσταση μόνο της Ρουμανίας, νομίζω και σε άλλες χώρες ενδέχεται να υπάρξουν φυσικές καταστροφές που να βάλουν σε κίνδυνο ένα πυρηνικό σταθμό. Την περασμένη εβδομάδα η Γερμανία πήρε μια απόφαση να μελετήσει το πώς παράγεται η ενέργεια. επιβάλλεται να αναθεωρήσουμε τα συστήματα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια μάλλον σε όλη την Ευρώπη και όλες οι χώρες πρέπει να έχουν αυστηρούς αυστηρότητους ελέγχους. Η Κομισιόν, η Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια να εφαρμόζεται σωστά. Επίσης η Κομισιόν από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να, ερευνήσει να εξετάσει τι συνθήκε σε όλου του πυρηνικού σταθμού. Η κατάσταση στην Ιαπωνία μα αποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων και των καταστροφών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκέρας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια για την Ιαπωνία. Πρώτα, καταρχήν πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ανακουφίσουμε τα βάσανα του Ιαπωνικού λαού που αξίζει κάθε υποστήριξη και συμπαράσταση από εμά. Δεύτερον, στην ε, τραγωδία του τσουνάμ και του σεισμού προστίθεται μια νέα τραγωδία του πυρηνικού σταθμού. Όλα αυτά μας οδηγούν σε μια πραγματική αλλαγή παραδείγματος, σε ένα σημείο τομής. Τι πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να ρωτήσουμε και δεύτερον τι μπορούμε να αλλάξουμε σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργεια στον κόσμο μας. Γιατί αν δεν υπήρχε ενέργεια από ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια, θα μπορούσαμε πολύ πιο νωρί να έχουμε καθορίσει μια στρατηγική για τι ανανεώσιμε ενέργειες. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαμορφώσει μια στρατηγική προ την κατεύθυνση αυτή. Χρειάζεται μια πολιτική θέληση και με ένα συγκεκριμένο φύλλο πορεία προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Έικχουτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και κυρία Ούτιγκερ. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ με την αρχή γιατί ξεκινήσατε γρήγορα την προηγούμενη εβδομάδα αλλά έκτοτε έχουμε καθυστερήσει και τώρα θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης χωρίς πυρηνική ενέργεια. Αυτό που το επαναλάβατε μετά από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή θα πρέπει να είναι η συζήτηση γιατί πολλέ έρευνες επιστημονικές καταδεικνύουν ότι μπορούμε να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους χωρίς πυρηνική ενέργεια. Μπορεί με βιώσιμη ενέργεια να ε, συνεχίσει η Ευρώπη. Είναι πολιτική αυτή η απόφαση αν υποστηρίξει κανείς την ε, πυρηνική ενέργεια ή όχι. Και δεν είμαστε εμείς που θα πρέπει να αμυνόμαστε ε, για, το τι, για τους λόγους για τους οποίους δεν θέλουμε ε, πριν η ενέργεια. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι δύο ερωτήσει. Έχω να σα κάνω, κύριε Ουτίνγκερ. Καταρχά, τι θα συμβεί, πώ θα ορίσουμε τα κριτήρια για να είναι ανεξάρτητα για τα stress test και τι θα γίνει αν ένα σταθμό δεν ε, πληρεί τα κριτήρια του stress test. Τι θα γίνει αυτό, ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Όλους μας λυπεί ιδιαίτερα η τραγωδία της Ιαπωνίας και θέλουμε να ποτίσουμε φοροτιμή τους ε, στα σωστικά συνεργεία που διακινδυνεύουν την ίδια τους τη ζωή για να ε, ανταπεξέλθουν στην κατάσταση μετά το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή. Αυτά που συνέβησαν στην ε, Ιαπωνία οδήγησαν σε μια έντονη συζήτηση στην Ευρώπη για το τι θα πρέπει να γίνει με την ενέργεια την ευρωπαϊκή. Προσφάτως, εγκρίναμε μια ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη για την περίοδο ως το 2020. Αυτή η στρατηγική πλέον φαίνεται ότι ε, τίθεται ένα αμφιβόλο. Στη στρατηγική αυτή αναφέρεται ότι η πρινική ενέργεια θα πρέπει να συνοδεύεται από πολύ αυστηρές ε, προδιαγραφές ασφάλειας, αλλά φαίνεται ότι αποτελεί ένα αποδεκτό τμήμα του ενεργειακού μείγματος κάποιων χωρών. Τώρα, έχω την αίσθηση ότι οι συζητήσεις μας θα πρέπει να κινηθούν προς την ε, κατεύθυνση της ενίσχυσης των όσων ε, ζητούμε στην έκθεση, δηλαδή πιο πολύ και πιο βαθιά ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα. Θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας ευρωπαϊκής ε, κοινότητας και αγοράς για την ενέργεια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πολιτική για την ενέργεια θα λάβει ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Τα stress οι δοκιμές αντοχές δεν θα πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση. Θα πρέπει να αποτελούν τμήμα της κοινή μας πολιτικής για την πυρηνική ενέργεια. Και πάνω απ' όλα θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες εδώ. Η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται στη διαφοροποίηση και στην αποκεντρώση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τους μικρούς πρινικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι στοιχίζουν λιγότερο, είναι πιο εύκολοι στον έλεγχο ασφάλειας. Ίσως αυτό να αποτελούσε μια πιο αποδεκτή λύση για τους ε, πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλτσίτης είναι επόμενος ομιλητής. Έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ιαπωνία <clears throat> έχει συγκλονιστεί από μια καταστροφή, μια φυσική καταστροφή χωρίς προηγούμενο. Ο λαός της Λιθουανίας συμπαραστέκεται στο λαό της Ιαπωνίας και συμμετέχει στην συλλογή αγαθών και χρημάτων για να βοηθηθεί η, η, η Ιαπωνία. <clears throat> Θυμόμαστε όλοι τα αποτελέσματα της πυρηνικής καταστροφής στο Τσερνομπίλ πριν από 25 χρόνια. Πρέπει όλα αυτά να μας οδηγήσουν να επανεξετάσουμε το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα ώστε οι φυσικές καταστροφές να μην επισύρουν περαιτέρω καταστροφές πιο σοβαρές όπως οι πυρηνικές καταστροφές. Όλα αυτά τα γεγονότα λοιπόν πρέπει να εξεταστούν και πάλι ιδίως μετά από την καταστροφή του Τσερνομπίλ που, ήταν ένα προηγούμενο. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που είναι απαραίτητο επομένω για να ενισχυθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η ποινική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντέιβι έχει το λόγο. Ένα λεπτό. <coughs> Χωρί μικρόφωνο, κύριο Ντέιβι. Εγώ ανησυχώ για την πυρηνική βιομηχανία, αλλά ανησυχώ περισσότερο για την κλιματική αλλαγή. Πιστεύω ότι η πυρηνική ενέργεια μπορούσε να μας βοηθήσει για τα θέματα αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης. Αυτό το πίστευα πριν από την κρίση στην Ιαπωνία και το πιστεύω ακόμα και τώρα. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ο σχεδιασμός των σταθμών, η σωστή ρύθμιση, δεν υπάρχει η απαραίτητη <clears throat> ανεξαρτησία των ρυθμιστών. Δεν μπορούμε να κάνουμε επίσης να κάνουμε ποινικού σταθμού σε σεισμογενείς ε, χώρους. Αλλά έχουμε ήδη πολλούς κινδύνους. Οι πόλεις μας είναι χημικά εργοστάσια. Πάρα πολύ ευαίσθητα. Τα καταφέρουμε. Είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα, τρομερά ατυχήματα με τρένα. Δεν έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε του ιδεοδρόμου. Μαθαίνουμε τα διδάγματά μα, τα εφαρμόσουμε και αυξάνουμε την ασφάλεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε και με την πυρηνική βιομηχανία. Κυρία Γιόρνταν Σίζελη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν όντω ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματο, η πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει τμήμα του ενεργειακού μείγματο δεν χρειαζόμαστε ιδεολογικές ε, ρητορίες. Πρέπει να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα πριν από αυτό. Και ποιος ήταν ο βασικός λόγος για το ατύχημα αυτό, πώς θα μπορούσε να έχει αποτραπεί. Υπήρχε ένα σύστημα εποπτείας το οποίο να λειτουργούσε. Υπήρχε ε, κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό. Πώς θα μπορούσαμε με καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας λειτουργούσαν σωστά οι ρυθμιστικές αρχές. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και μόνο τότε μπορούμε να αναλάβουμε πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική συμφωνία για το ποιε ποιες τεχνολογίες είναι αποδεκτές. Συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής τεχνολογίας θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή ότι πρώτα απ' όλα έρχεται η ασφάλεια. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε να ορίσουμε το αριθμιστικό πλαίσιο με την απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο εργατικό δυναμικό για θέματα ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη, να είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και να υπάρχει και μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ των γενεών. Επίσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι ρυθμιστικές αρχές είναι επαρκώς ανεξάρτητες και επίσης να φροντίσουμε για την ασφαλή απόρριψη των αποβλήτων. Ολοκληρώνοντας, υπάρχουν κάποια κοινά κριτήρια ασφάλειας και όλοι σήμερα γνωρίζουμε ότι τα χρειαζόμαστε αυτά τα κοινά κριτήρια. Το 2009, όταν συζητήσαμε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τέτοια κριτήρια και δυστυχώς το Συμβούλιο δεν τα αποδέχτηκε τότε. Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει πιο πολλές αρμοδιότητες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και θα πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συμφωνίες στα πλαίσια της συναπόφασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λιμπεράτσκι είναι στον κατάλογο, δεν τον βλέπω όμως, δεν είναι παρόν. Ωραία. Και έτσι θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Γκόλ Πέλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να εκφράσω την, ε, τα συλληπιτήριά μου προς τον λαό της Ιαπωνίας και επενώ το κουράγιο τους, το θάρρος τους, την αποφασιστικότητα τους αυτών των ε, ηρώων που σήμερα αγωνίζονται ενάντια στην πυρηνική καταστροφή. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα θυμόμαστε σε όλη μας την ιστορία. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν συντονισμένη και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε άμεσα και επανέλαβε ότι το μισό εκατομμύριο κόσμος που επλήγησε από το σεισμό και το τσουνάμι θα λάβει βοήθεια. Πέραν όμως αυτών, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουμε τέτοιες συμφορές, τέτοιες καταστροφές και για να βοηθήσουμε το λαό της Ιαπωνίας να ξαναμπεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Τέτοιας έκτασης καταστροφές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα κατά της πυρηνικής ενέργειας. Αντιθέτως, τα πυρηνικά εργοστάσια θα πρέπει να υπόκειται στις πιο αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και να, συνεχί... να βρίσκονται υποδιαρκή ε, έλεγχο. Θα πρέπει να γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις και είμαι υπέρ των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα κατατεθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα παρέχουν μια συντονισμένη βάση για την ασφάλεια και θα εγγυηθούν την ασφάλεια στο μέλλον της ενεργειακής, ε, της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι θα... Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Εντίτ Χερτσόγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συναδελφοί. Σήμερα όλοι είμαστε Ιαπωνέζοι, εν μέρη. Ακόμα και μπροστά σε θεομηνίες θα πρέπει να δούμε ένα, ένα ανθρώπινο πρόσωπο για την πυρηνική ασφάλεια, προγραμματισμός, λειτουργία και κλείσιμο του σταθμού. Όλα αυτά τα, ε, ε, τα διαχειρίζονται άνθρωποι. Και ζώντας στην καταστροφή βλέπουμε το πρόβλημα για τους ανθρώπους. Το τεστ κόπωσης είναι σημαντικό βήμα βέβαια. Πρέπει να προγραμματίσουμε για απρόβλεπτα γεγονότα στο μέλλον. Κύριε Πίτροπε, Πρέπει να εκφράσουμε το σεβασμό μας για την δουλειά που γίνεται στη Φουκοσίμα. Πρέπει οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες να πάρουν μέρος στην επεξεργασία πολιτικής. Αυτοί που δουλεύουν στα πυρηνικά εργοστάσια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη τους, τις γνώσεις τους. Μεσοπρόθεσμα χρειαζόμαστε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη γιατί αυτό είναι εγγύηση για πυρηνική ασφάλεια. Και ευχαριστώ την προσοχή σας το κάτι που ανέφερε και ένας άλλος συνάδελφος. Η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να δώσει καλύτερες απαντήσεις στο πώς θα χειριστούμε τα πυρηνικά απόβλητα από εδώ και μπρος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε στη διαδικασία Catch the Έχουμε ένα πρόβλημα γιατί έχω 15 άτομα στον κατάλογο και έχω μόνο 5 λεπτά. Θα πάρω 6 συναδέλφους. Θα διαιρέσω ισότιμα ε, το χρόνο με βάση τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Ρούμπικ πράγματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο Έτουγκερ γιατί έδειξε πνεύμα υπευθυνότητος για το ζήτημα αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε αν θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση των πυρηνικών σταθμών και με ποιο τρόπο, αν θα πρέπει να γίνει από τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν οι κανόνες μας θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί και αν δεν τηρούνται τα πρότυπα θα έχουν οι νέε ρυθμιστικές αρχές να κλείνουν τους πυρηνικούς σταθμούς. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και για μια μεταρρύθμιση της συνθήκης Ευρατόμ όπου να δίνουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών και επίση για τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για το κλείσιμο των ποινικών σταθμών και την οριστική απόθεση των αποβλήτων. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν και τη δυνατότητα στην Ευρώπη να υπάρχει ένας έλεγχος ομοτήμων για τα νέα αυτά πρότυπα ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Κύριος Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά Καλωσορίζω την ε, γοργή αρρωγή προς τους Ιάπωνες και καλωσορίζω και τη συμπάθεια που εκφράζουμε προς τους Ιάπωνες. Ωστόσο, αναρωτιέμαι για το κατά πόσο είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε για αλληλεγγύη και μήπως αυτό επηρεάζεται από κάποιες δράσεις των κρατών μελών. Διαβάζοντας τις εφημερίδες βλέπουμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση ελέγχει για ακτινοβολία τα τρόφιμα από την Ιαπωνία, ότι η Ολλανδική κυβέρνηση ε, και οι γερμανικές αρχές, οι γαλλικές αρχές ελέγχουν όλες ε, τις εισαγωγές και τα αυτοκίνητα ακόμα. Πρόεδρε, αυτά συμβαίνουν δύο-τρει εβδομάδε μετά τον σεισμό. Είναι περιορισμένη η έκφραση αλληλεγγύη σε τέτοιε δράσει. Ζητώ από την Κομισιόν και στο Συμβούλιο να μιλήσουν με τα κράτη-μέλη για να μην ε, ε, ακούγονται τέτοιε ιστορίε τρόμου. Ευχαριστώ κυρία Χώρη, στην επόμενη ομιλητρία. Μου προκαλεί έκπληξη που φαίνεται τόσο αισιόδοξο ο επίτροπο για το ότι θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την κατάσταση στη Φουκουσίμα μέσα σε λίγες ημέρες, όταν οι εμπειρογνώμονες μιλούν για εβδομάδες και για μήνες και μεταξύ εξακολουθεί να εκπέμπει ε, ραδιενέργεια η, ο σταθμός Καλωσορίζω τα stress test, αλλά δεν απαντούν τα μεγαλύτερα ερωτήματα που τίθενται. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να αποδεχτούμε τον ολοένα και αυξανόμενο κίνδυνο των πυρηνικών εργοστασίων σε έναν κόσμο όπου οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται διαρκώς. Η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων πολύ απλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε απόλυτα να εγγυηθούμε σε περίπτωση μιας μεγάλης ε, καταστροφής οποιαδήποτε φύσεως. Είτε υπάρχουν πολλά ε, επίπεδα καταστροφής όπου υπάρχουν ε, για παράδειγμα διακοπές ηλεκτρικού και νερού ή πρόσβασης ή προβλήματα πρόσβασης. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα. Θέλουμε να πάρουμε αυτό το κίνδυνο όταν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να εκφράσουμε όλοι μας τη συμπαράσταση και την αλληλική μας προς το λαό της Ιαπωνίας και δίνουμε και τα δικά μας συλληπιτήρια προς τους οικείους των θυμάτων της καταστροφής. Αυτή η καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα έχει συνέπειες οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί σε όλη την έκτασή τους. Έγινε αυτό το οποίο ήταν πραγματικά απίθανο. Είναι γεγονός αλλά αυτό δείχνει ότι μπορεί κάτι τέτοιο να επαναληφθεί σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς. Γι' αυτό πρέπει να αντλήσουμε σημαντικά διδάγματα για αυτό το οποίο έγινε στη Φουκουσίμα. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας των ε, πυρηνικών σταθμών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα ψήξης. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την ε, τοποθεσία τον ε, πυρηνικό σταθμό σε σχέση με τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών και ιδίω σεισμού. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε και μια ευρεία συζήτηση στην κοινωνία μα για την ενεργειακή μα πολιτική στο μέλλον και για τον τρόπο με τον οποίο θα ικανοποιηθούν οι ενεργειακέ μα ανάγκε. Με έναν τρόπο ο οποίο θα είναι διαυγή και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι δυνητικέ επιπτώσει για τι ε, πηγέ ενέργεια που μπορούμε να επιλέξουμε. Κύριος Ρώση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν συμφράσουμε την αγγελική μας στον Ιαπωνικό λαό που επήγε από την καταστροφή αυτή. Ήταν έκπληξη η Ιαπωνέζικη τεχνολογία να βρεθεί off-site σε μια περιοχή μάλιστα που συμβαίνουν ένα σωρό σεισμοί. Το να κρατήσουν σε εμπειρικό σώμα σε λειτουργία ενώ είναι τεχνολογικά ξεπερασμένου σίγουρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σημείο. Και αυτά όλα θα πρέπει να μα κάνουν να σκεφτούμε το ευρωπαϊκό πυρηνικό πρόγραμμα μην αφήσουμε να μας κυριαρχήσει ο φόβος σήμερα. Χρειάζεται γενική συμφωνία για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και ένα screening για αυτούς που θα κατασκευαστούν εφ' εξής. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να επενέσουμε και να παρακολουθούμε το τι έγινε στην Ιαπωνία γιατί μπορεί να έχει, να έχει και συνέπειες σε άλλες μορφές κρίσης. Μπορεί να επιβαρυνθεί η οικονομία και χώρε που συνδέονται με την Ιαπωνία να υποστούν τον αντίκτυπο. Μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ήδη και πριν την καταστροφή ήταν ασθενή και χωρί πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα ε, υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει η κυβέρνηση. Πρόεδρος, η Αγγέλικα Βέρτμαν. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχά να πω ότι συμπάσχω με όλους του από την τραγική αυτή καταστροφή. Το τραγικό ατύχημα μας οδήγησε στις, ε, σε μια χωρική αντίδραση στην Ευρώπη. Ωστόσο, συνειδητοποιούμε τουλάχιστον σε όλους τους προσασπιστές της ε, πυρηνικής ενέργειας ότι δεν υπάρχουν όρια στην ραδιενέργεια. Ούτε η φύση έχει πρότυπα ασφαλείας. Στο Τσέρνομπιλ ήταν ένα αποτυχημένο στρες τεστ και έχουμε τώρα και την ε, Φοκουσίμα. Είναι καιρός πια οι προασπιστές της πυρηνικής ενέργειας να θέσουν την ευημερία και την υγεία του ανθρώπου πάνω από όλα. Να σκεφτούμε λοιπόν ε, μια ευρωπαϊκή αποχώρηση από την πυρηνική ενέργεια. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ιαπωνία επλήγει από ένα τσουνάμι μετά από ένα σεισμό που οδήγησε σε μια πυρηνική καταστροφή. Η πυρηνική καταστροφή θέτει το θέμα της ασφάλειας του πληθυσμού και των εργαζομένων στους πυρηνικούς σταθμούς. Όλα αυτά μας οδήγησαν στα stress test γιατί είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια πλήρη συζήτηση για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστά πληροφορημένη απόφαση για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι μετά από μια τραγωδία αυτού του μεγέθους θα υπάρχει μεγαλύτερος φόβος στην κοινή γνώμη. Πρέπει να είμαστε πάρα προσεκτικοί για να δώσουμε αντικειμενική αλλά και σαφή πληροφόρηση στον πληθυσμό σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Θέλω να τονίσω ότι οι κλιματικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν κινδυνεύει από τσουνάμι, ούτε τόσο έντονους σεισμούς. Επομένως δεν μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα άμεσα από αυτή την τραγωδία σε σχέση με τους κινδύνους στην Ευρώπη η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει και τμήμα του ενεργειακού μας μίγματος στο μέλλον και φυσικά θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήρια προς τους Ιάπωνες φίλους μας. <clears throat> Ερχόμαστε τώρα στην ε, ε, απάντηση του κυρίου Επιτρόπου και του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω ακούσει με μεγάλη προσοχή τις παρατηρήσεις των ε, βουλευτών και νομίζω ότι υπήρξε μια μεγάλη ικανότητα σε επίπεδο αντικειμενικότητας και γνώσης των πραγμάτων και μια νυφαλιότητα σε σχέση με τις συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Από την πλευρά του Συμβουλίου και της Κομισιόν έχουμε προβλέψει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στην ε, ασφάλεια σε γενικό επίπεδο. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καταστροφών τα πρόσφατα χρόνια. Η ΑΕΤ, το Πακιστάν, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις <clears throat> η Κομισιόν είναι αυτή η οποία είναι αρμόδια για να αξιολογήσει το μέγεθος της καταστροφής και το Συμβούλιο θέτει τις πολιτικές κατευθύνσεις πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αντιμετώπιση καταστροφών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά και ανθρώπινα μέσα στη διάθεσή μας και φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε έμφαση στον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας. Και η Κομισιόν είναι έτοιμη να θέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα συμπράσματα που πρέπει να αντλήσουμε από την καταστροφή της Φουκουσίμα και τις συνέπειες για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα και την πραγματικότητα με έναν τρόπο ο οποίος είναι αντικειμενικός και σαφής. Η γερμανική κυβέρνηση ε, στην οποία συμμετέχει και ένα κόμμα το οποίο προέρχομαι εγώ, έχει προβεί σε μια σημαντική στροφή. Ε, έκλεισε προσωρινά 7 ποινικού σταθμούς και η απάντηση ήταν το άγχος, ο φόβος στη Γερμανία. Εγώ πιστεύω όμως ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε το σεβασμό και για την αντίθετη θέση. Εγώ έχω μεγάλο σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έδωσε την έγκρισή του στο να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και ποινική ενέργεια. Εγώ έχω απόλυτη, επίσης, απόλυτο σεβασμό για τις ρυθμιστικές αρχές και την ικανότητά τους και τις αρχές της Ευρατόμ και επίση και για τι αρχέ ασφαλεία, οι οποίε ενεκρίθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέλαβαν τα καθήκοντα του πριν από δύο χρόνια. Υπήρξαν πολλέ ενέργειε σε επίπεδο τυπικό, δηλαδή για τις αρχές της ίδιας, για, το, για την υποχρέωση να παρέχουν ε, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και επίσης συγκεκριμένες προδιαγραφές σε επίπεδο κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών πυρηνικής ενέργειας. Αν εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλετε να επεκτείνετε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα θέματα αυτά, δεν θα πρέπει να αναμένουμε μόνο τις <clears throat> εκθέσεις των κρατών μελών τα επόμενα δύο-τρία χρόνια, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μία εξασφάλιση ότι θα υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν στη συνέχεια στο εθνικό δίκαιο και με τη βοήθεια των εμπειρογνωμοσυνών από την Ιαπωνία και των stress test θα μας οδηγήσουν σε περαιτέρω προτάσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών και οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εγώ θέλω να φανώ συνεπής και να, να ακολουθήσουν τα θεσμικά όργανα τις αρμοδιότητες που έχουν Εγώ έτυχα επικρίσεων από εθνικές κυβερνήσεις για το γεγονός ότι εγώ έκανα μια κάπως ρηξικέλευτη αξιολόγηση της κατάστασης στη, Φου, στη Φουκουσίμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις αρμοδιότητες που έχουμε. Και θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι όταν έχουμε 153 πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη και όταν έχουμε αυτούς τους σταθμούς οι οποίοι θα παραμείνουν την επόμενη δεκαετία και ίσως θα υπάρξουν και περισσότεροι σταθμοί οι οποίοι θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στην Ευρώπη τότε το συμφέρον της Ευρώπης, το συμφέρον όλων μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα Ποινικά αυτά εργοστάσια που θα λειτουργούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα ανταποκρίνονται σε, υψηλά, σε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια όλων. Δεύτερον, θεωρώ ότι για την Ευρώπη το θέμα της κατασκευής περαιτέρω ποινικών σταθμών είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινοβουλίων τους. Υπάρχει ένα δημοψήφισμα το οποίο θα λάβει η χώρα στην Ιταλία το καλοκαίρι προς την κατεύθυνση αυτή και στην, σε καμία από τις 13 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πυρηνικούς σταθμούς δεν υπήρξε με την εξαίρεση της Γερμανίας καμία απόλυτη αλλαγή της κατεύθυνσης. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε στην Ευρώπη και μία ακόμα ε, μία άλλη διάσταση. Σε παγκόσμιο επίπεδο θα εξακολουθήσουν και έξω από την Ευρώπη να υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί. Δεν θέλουμε πρότυπα μόνο για μας, θέλουμε πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς διακόπτη ο κύριος Τούρμες χωρίς, χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Τούρμες. Όταν λέτε ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη σε μας, εγώ έχω εμπιστοσύνη γιατί το θέμα αυτό έχει έρθει ότι θα έρθει το θέμα αυτό στη μέση διάταξη των G20 όπου και οι Αμερικανοί και άλλες χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικούς σταθμούς και οι χώρε οι οποίε έχουν μεγάλε επιχειρήσει, οι οποίε δημιουργούν πυρηνικού σταθμού, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εκ νέου αξιολόγηση των κινδύνων και των προτύπων ασφαλεία είναι απαραίτητη. Ακόμα είτε κανείς υποστηρίζει την πυρηνική ενέργεια είτε είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί η πυρηνική ενέργεια, κυρία Χάρμς πάλι χωρίς μικρόφωνο, Αφήστε τον, τον ε, ομιλητή να, να περατώσει. Δεν, πρέπει να έχουμε μία ε, λανθασμένη αντιμετώπιση. Εγώ νομίζω ότι αυτή η οπτική που ακολουθεί η Κομισιόν είναι η σωστή σε αυτά τα θέματα. Και η στόχοι του 2050 το ότι δεν θα επαρκέσουν οι οι χρηματοδοτήσει για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Εδώ εσείς υποτιμάτε ήδη τις αποφάσει που έχετε λάβει εσεί ήδη. Το 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα επόμενα 9 χρόνια, αυτό σημαίνει για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35%. Αν το 35% του ρεύματος μπορεί να παράγεται από ανανεώσιμες ενέργειες, τότε αυτό θα σημαίνει ότι σε τέσσερα χρόνια, ότι σε πέντε χρόνια μπορούμε να ανακτήσουμε το τμήμα αυτό της παραγωγής το οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε μάλλον την πυρηνική ενέργεια σε ποσοστό παραγωγής και να ξεπεράσουμε και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον άνθρακα. Θα είναι οι ανανεώσιμες ενέργειες το σημαντικότερο τμήμα της ε, παραγωγής ενέργειας. Έτσι θα είναι το σημαντικότερο τμήμα της, ε, του σενάριου που θα ακολουθήσουμε. Αλλά αυτό ε, δεν αφορά μονάχα το 2050, αφορά το 2025, το 2030, την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, την απαραίτητη δυνατότητα ε, παραγωγής ενέργειας, θα πρέπει να επενδύσουμε σε όλες αυτές τις πτυχές. Το 2030 δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο 35% ανανεώσιμης ενέργειας, θα πρέπει να έχουμε 40% και περισσότερο. Μπορεί το 40% να είναι ο μέσος όρος ή ακόμα και περισσότερο αυτού. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε δεν θα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν υποστηριχθεί αρκετά οι ανανεώσιμες ενέργειες, αλλά ότι έχουμε καταφέρει να είναι το αποφασιστικό κομμάτι του ενεργειακού μείγματος για ανανεώσιμες ενέργειες. Εκτός, Εκτός μικροφώνου, κύριε Χάραμς. Κύριε μιλώ για τον οδικό χάρτη της ενέργειας. Εσείς μιλάτε για τα θέματα διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι όμως το ίδιο αυτό, ξέρετε. Δεν είναι το ίδιο, λέει ο Επιτρόπος. Έχουμε τους στόχους για το 2020. Το αφήσατε στο 20% τους στόχους και 30% αυτό αποφάσισαν Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν και αυτό προτάθηκε. Καμία αλλαγή. Τώρα όμως μιλάμε για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Εδώ θα ξεπεράσουμε το 40%. Δημιουργήσαμε μία βάση προκειμένου αφενός το ενεργειακό μείγμα να μην είναι μόνο θέμα των κρατών μελών, σε καμία περίπτωση τα κράτη-μέλη κατά 50% ή και κάτι παραπάνω ε, έχουν αρμοδιότητα και κατά δεύτερον δώσαμε προδιαγραφές για το πώς ε, θα πρέπει να είναι η βάση ενίσχυσης ε, οικονομικά και τεχνικά στα κράτη-μέλη. Και μπορείτε να θεωρήσετε ότι στα σενάρια ε, συνάδελφε Τούρμες, ε, ε, ελέγχεται ένα πράγμα. Από διάφορες ενώσεις έχει προταθεί αυτό. Το σκοπός μας είναι να πάμε στο 100% ανανεώσιμες ενέργειες. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε το άρθρο 194, όπου αναφέρεται ότι το ενεργειακό μείγμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και θεωρώ ότι δεν είναι η βίβλος η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά αποτελεί, εν περιπτώσει, τη βάση της δουλειάς μου. Και θα πρέπει να σέβομαι τα δικαιώματα των κρατών μελών, ούτε είτε είναι η Ιταλία, το, ε, το Λουξεμβούργο, το Λονδίνο κτλ. Τελευταίο σημείο. Άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι Ντέιβις και Χαλ και οι δύο στο ίδιο κόμμα ανήκουν και ιδίω σε ένα κράτος μέλος και οι δύο με εντελώς αντίθετη άποψη. Τη σέβομαι την άποψη αυτή, αλλά όταν ένα μικρό κόμμα σε μια μεγάλη χώρα είναι τόσο διχασμένο, και αυτό φαίνεται από δύο αξιότιμους βουλευτές, και το ίδιο κόμμα πριν από τις εκλογές ήταν κατά των πρινικών εργοστασίων και μετά τις εκλογές ε, έκανε, τα τακτοποίησε και έκανε συμβιβασμούς αυτό δείχνει τη διάσταση οικολογικής, οικονομικής και οικονομικής διάστασης. Πόσο περίπλοκη είναι η διαδικασία αυτή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Επιτρόπε λέει ο πρόεδρος, η κυρία Γκέρι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κυρίε και κύριοι, θα είμαι σύντομη. Νομίζω πρέπει να δείξουμε την συμπαράστασή μα και ψυχραιμία για να μπορέσουμε να δράσουμε. Πρέπει να δράσουμε τα συλληπιτήριά μας, να δώσουμε βοήθεια στους Ιαπωνέζου, να του δώσουμε ό,τι χρειάζονται να του ακούσουμε, να είμαστε παρόντε εκεί αν μα χρειαστούν και χρειαζόμαστε και ψυχραιμία για να σκεφτούμε το μέλλον και να πάρουμε τις αναγκαίες αποφάσεις. Δεν πρέπει να βιαστούμε λόγω των σημερινών γεγονότων και να πάρουμε λάθος αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι εδώ μέσα συμφωνούμε με αυτό. Ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, εσωτερική και εξωτερική. Επίσης να πληροφορήσουμε τους πολίτες μας πλήρως για να καταλάβουν πώς έχει η κατάσταση και τι θα κάνουμε, πότε και πώς. Εξίσου σημαντικό είναι να διδαχθούμε από τις συνέπειες, να αναλύσουμε την κατάσταση γρήγορα, χωρίς όμως να προδικάσουμε τίποτα και χωρίς να κάνουμε δηλώσεις οι οποίες μετά από μερικές εβδομάδες ή μήνες δεν μην ισχύουν. Όσον αφορά τα τεστ κόπωσης, με βάση το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο ε, είναι δυνατόν να γίνουν προαιρετικά. Πολλοί από εσάς είπατε, νομίζω και το Συμβούλιο θέλει να αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο του ισχύων. Χρειάζονται όμως προτάσεις. Χρειάζονται να συζητηθούν οι προτάσεις, όχι βιαστικά. Πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά. Ο κύριος Επίτροπος ανάφερε επίσης το μείγμα ενεργειών. Αυτό είναι θέμα εθνικό. Κάθε χώρα το αποφασίζει. Τι είδους πηγές ενέργειας θα ενσωματώσει σε αυτό το ενεργειακό μείγμα. Περίπου οι μισές χώρες μέλη χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούμε να ορίσουμε κανόνες για την ασφάλεια την ευθύνη την έχουν, μάλλον ό,τι και να κάνουμε, την ευθύνη τελικά την έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Και ε, επισημαίνω ιδιαίτερα θετικά το ότι ο Επίτροπος για την έκθεση αυτή είπε ότι θα είναι έτοιμη μέχρι τον Ιούλιο. Μία τελευταία ιδέα τέλος είναι η έρευνα και η ανάπτυξη. Το συζητήσαμε πολύ στα πλαίσια της στρατηγικής 2022, γιατί είναι ο ένας από τους αυτής της πολιτικής η έρευνα και η ανάπτυξη πρέπει να ε, έχει τις, τους καλύτερους δυνατούς όρους στην Ένωση. Πρέπει να έχουμε την πιο, τις πιο ασφαλείς μορφές, μορφές παραγωγής ενέργειας, τις πιο αποδοτικές. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την επιστήμη προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη ασφάλεια για τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κυρία Γιώρη. Περατώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό, η ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Το επόμενο θέμα είναι η προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για ένα κοινό πρόγραμμα